Alliance και αυτά θα καταγραφούν και στα πρακτικά της τρέχουσας συνόδου. Ερχόμαστε τώρα στην για διάταξη, η οποία έχει αποφασιστεί από την συνέλευση των Πρόεδρων στις 20 Μαρτίου στην οριστική της μορφή και έχει διανεμηθεί στους βουλευτές. Εγώ προτείνω σε σχέση μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες η έκθεση της κυρίας Βίξτρομ για την προστασία της ε, ασυλίας του κυρίου Βλάντιμ Τουντόρ να περιληφθεί κατευθείαν στον χρόνο των ψηφοφοριών. Και έτσι έχουμε ε, εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη ανησυχία σας πληροφορώ για τα τελευταία γεγονότα στο Μπαχράιν υπήρξε μεγάλη πίεση για καταστολή κατά αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει οξυνθεί τι τελευταίε μέρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την κυβέρνηση του Μπαχρέν, εξονόμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την υποχρέωσή τη να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι συμφωνίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν ηθική και υλική δέσμευση για την κυβέρνηση του Μπαχρέν και κατ' ό,τι η κυβέρνηση του Μπαχρέν να έρθει σε επαφή με όλε τι πολιτικέ δυνάμει στην χώρα αυτή. Επίσης, θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Και στην Αίγυπτο η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Δεν είναι δυνατόν μετά από ένα χρόνο μετά από την ανατροπή του Μουμπάρεκ να εξακολουθεί να υπάρχει καταστολή κατά συγγραφέων blog, ε, πολιτικών σχολιαστών κτλ. Εξακολουθεί η δίκη κατά του Ασμάρ Μαχμούς ο οποίο έχει πάρει το βραβείο Σαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί ω Κοινοβούλιο θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πλευρά όλων αυτών, οι οποίοι στι γειτονικέ μα χώρε ή και σε άλλε περιοχέ του κόσμου εξακολουθούν να αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την πλουραλιστική και ανεκτική κοινωνία που θέλουμε να έχουμε. Και εδώ θέλω να φέρω και την περίπτωση του κ. Βεντζεσλά Μανζόγκο στην Ισημερινή Ουινέα, ο οποίο και αυτό είναι αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα θέλω να εκφράσω την θλίψη όλων μας για το θάνατο ενός αγαπητού συναδέλφου, του Μιγγέλ Σακαντούρα Πόρτας, ο οποίος